Να σας ανακοινώσω επίσης ότι σέλαβα από την ομάδα των Ελευθέρων Δημοκρατών και Φιλελευθέρων για την Ευρώπη ο εξή στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας η κυρία Σιλβάνα Κοχμερίν γίνεται τακτικό μέλος ε, και αντικαθιστά τον ε, κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη. Τελευταία ανακοίνωση.